κοινωνίας των πολιτών ε, και διάλογος έχουν ήδη ξεκινήσει με το Περού αλλά και με άλλες χώρες για το θέμα της μπανάνας. Όπως γνωρίζετε, οι όροι για την προσωρινή άρση εφαρμογής των προτιμήσεων περιλαμβάνονται ήδη στην συμφωνία, χωρίς όμως αναυτοπαντοποιημένη απόφαση. Αυτό έχει να κάνει, θα εξαρτηθεί από μια αξιολόγηση της σταθερότητα της αγοράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάθε φορά λοιπόν που υπάρχει αυτή η υπέρβαση επίπεδο Λατίνική Αμερική, όπως έγινε και πέρυσι, εμείς από πλευράς Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέβημε σε μια ει βάθος ανάλυση, καταλήγοντα στο συμπέρασμα ότι η υπερ υπερβολικές εισαγωγές δεν αποσταθεροποιούν τις ευρωπαϊκές αγορές και έχουν μικρή επίπτωση στην διαμόρφωση των τιμών της μπανάνας. Ωστόσο, συνεχίζουμε την παρακολούθηση του θέματος. Στις ε, κατεψυγμένες ε, τηγανιτές πατάτες ε, που επισήμανε ο Βέλγος συνάδελφος, βεβαίως και είμαστε εν γνώση του θέματος, το έχουμε επισημάνει στις αρχές Κολομβίας επανελειμμένως, συμμερίζομαι και εγώ τις ανησυχίες σας. Έχουμε βέβαια κάποιο πρόβλημα σε σχέση με τον τρόπο υπολογισμού των μεγεθών. Με την Μπογκοτά λοιπόν την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε συνομιλίες η ομάδα δηλαδή των εμπορικών συνολεγών των αρχών της Κολομβίας ε, θα είναι παρούσα και θα συζητήσουμε μαζί τους στην Πογκοτά για τα θέματα αυτά και θα σας ενημερώσουμε για περαιτέρω εξελίξεις. Όπως είπα έχουμε ξεκινήσει μια συνολική αξιολόγηση των δύο αυτών συμφωνιών. Πολύ ευχαριστώ θα σας ενημερώσουμε μόλις ολοκληρωθεί για να ξανασυζητήσουμε τα θέματα αυτά σε μεταγενέστερο στάδιο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα οι δύο τελευταίοι ομιλητές, οι συγητές, ο κύριος Φίσας Αουξέρα. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επίτροπο Μάλστρομ και όλους τους συναδέλφους για τις ενδιαφέρουσες ομιλίες τους και τη συνεισφορά τους απόψε. Είναι φίλη η περιφέρεια η Λατινική Αμερική. Έχουμε πολύ ισχυρού ιστορικούς δεσμούς μαζί της και οι ε, τελευταίες εμπορικές συμφωνίες ενισχύουν αυτή τη σχέση και δίνουν και μια προοπτική ε, της ε, στρατηγικής και γεωπολιτικής σημασίας που έχει η Λατινική Αμερική για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αγαπητέ φίλε Χέλμουτ, σε τιμώ, αλλά θα πρέπει να καταλάβουμε ε, και να εκτιμήσουμε από πού έρχονται και πού έχουν φτάσει τώρα αυτές οι συμφωνίες ε, και οι χώρες. Το να ανασταλούν οι συμφωνίες θα ήταν το χειρότερο που θα μπορούσαμε να κάνουμε, όπως είπε και ο Ραμόν Χάορεγγι. Και αγαπητέ Γκαμπριέλ και ε, άλλοι συνάδελφοι, ε, ε, θα πρέπει να προσέξουμε τα θέματα της μπανάνας, ε, τα είπε και η Επίτροπος. Το Περού και η Κολομβία και ο Ισημερινός είναι στρατηγικέ περιοχέ για την Ευρωπαϊκή Ένωση, άρα έχει απόλυτη σημασία να συνεχίσουμε να προωθούμε τι ε, συμφωνίε αυτέ για να αναπτύξει το πλήρε δυναμικό τη. Και θυμίζω ότι υπάρχει και μια ρήτρα προσχώρηση. αφήνει ανοιχτή την πόρτα έτσι ώστε να συμμετάσχουν και άλλα ε, μέλη ε, της κοινότητας των Άνδεων, χώρες της περιοχής. Δεν θα ήθελα να τελειώσω την παρέμβασή μου χωρίς να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους από την Επιτροπή Ίντα και ιδιαίτερα τους κοιόδη ηγητές και τη συνάδελφο Ροντρίγε Πινέιρο κυρίως ε, που μα βοήθησαν να φτάσουμε σε μια έκθεση ισόρροπη, θετική και ελπίζω αύριο να υπερψηφιστεί με πολύ μεγάλη υποστήριξη στην Ολομέλη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Και τώρα το λόγο έχει ο κύριος Ράιμερ Μπέγκε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ευθύς εξ αρχής, δεδομένης ε, της κριτικής, της δικαιολογημένης και των παρατηρήσεων που ακούσαμε. Εκκρεμούν ακόμα πολλά θέματα ε, στις σχέσεις μας με τις εταιρικέ αυτές χώρες. Θα πρέπει να προχωρήσουμε και με πίεση αλλά και με σύνεση και μέτρο Κυρία Επίτροπε, εσεί πραγματικά τα τελευταία χρόνια έχετε επιτελέσει ένα πολύ σπουδαίο έργο στην ε, εμπορική πολιτική. Θα πρέπει να πω στου συναδέλφου ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε, όπω είπε και ο κύριο Φίσα, από πού ε, ξεκίνησαν οι χώρε αυτέ, και να μην απαιτούμε το 100% την απόλυτη εφαρμογή τη συμφωνία, αλλά να το δούμε δυναμικά. Ποιε είναι οι πρόοδοι και πώ έχει προχωρήσει η συμφωνία. Και έρχομαι σε ένα άλλο θέμα τώρα, κύριε Πρόεδρε. Κοιτώντα τι χώρες για τις οποίε συζητήσαμε εδώ Περού και Κολομβία. 500.000 ε, πρόσφυγες έχει και μόνο το Περού υποδεχτεί και η Κολομβία ένα εκατομμύριο από τη Βενεζουέλα. Και οι χώρες αυτές είναι σε μια ευαίσθητη εύθραυση κατάσταση, σχεδόν στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Εμείς κάνουμε αρκετά ε, ε, μαζί με την είπατε αρμοστία το ΟΗΕ για τους πρόσφυγες ή εξακολουθούμε να μην κάνουμε αρκετά. Ε, έχουμε πραγματικά ένα διαολεμένο καθήκον ως Ευρωπαϊκή Ένωση να δράσουμε και με όλη τη γειτονική περιοχή της Λατινικής Αμερικής για να μην δηλητηριαστεί και να μην καταστραφεί. Γιατί από τη μια μέρα στην άλλη θα καταρρεύσουν όλες οι προσπάθειες, όχι μόνο στην εμπορική πολιτική, θα πρέπει παντού να εφαρμόζονται αυτά που ζητούμε. Και δεδομένης και της αλαζονίας των Ηνωμένων Πολιτικών και της καταγγελίας της συμφωνίας με τον Ειρηνικό, εμείς δεν θα πρέπει να σταυρώσουμε τα χέρια και να αφήσουμε έρμεο στα χέρια ε, άλλων μεγάλων δυνάμεων όπως είναι η Κίνα την περιοχή αυτή, στην αλαζονία και την περιφρόνηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Όλα αυτά θα πρέπει να μας απασχολήσουν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει και ο Πρόεδρος, ε, ε, τον εισηγητή μας, τον κύριο Μπέργκε. Ολοκληρώνεται εδώ η κοινή συζήτηση. Η ψηφοφορία θα γίνει αύριο. Προχωρούμε στο επόμενο θέμα κατά την ημέρησια διάταξη, αλλά έχουμε μια ανακοίνωση ο κύριος Ινελίνε φεύγει από το ΕΛ και προσχωρεί στην ομάδα του ECR, των συντηρητικών και μεταρρυθμίσεων από αύριο. Η κυρία Τζέιν Κόλλινς και ο κύριος Τζον Στουαρτ Άντνιου αποχωρούν από την ομάδα EFTD και προσχωρούν στην ομάδα ENF από αύριο, 16ης πρώτου. Ο κύριος Τζέραλτ Μπάττον πάβει να είναι μη εγγεγραμμένος και εντάσσεται στην ομάδα ENF από τι 16 Πρώτου 2019. Αυτέ ήταν οι δηλώσει που είχα να σα κάνω και ανακοινώσει και προχωρούμε στο επόμενο θέμα τη ημερήσια διάταξη, που είναι η έκθεση κυρία Μαρία Ρενά, Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Θα θέλαμε να καλωσορίσουμε και την Επίτροπο Τάισεν και όλους συμμετέχοντες σε αυτή τη συζήτηση. Κυρία Ρένα, έχετε το λόγο ως εισηγήτρια. Ευχαριστώ, ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ κυρία Επίτροπε. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Παγκοσμιοποίηση που δημιουργήθηκε το 2006 είναι ένα ταμείο αλληλεγγύης και βοηθάει τους εργαζόμενους που είναι θύματα αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων μετά την παγκοσμιοποίηση. Εδώ και 10 χρόνια αυτό το ταμείο παρακολούθησε 150.000 εργαζόμενους μέσα στα πλαίσια 150 επιχειρήσεων υπό αναδιάρθρωση και έχουμε και 4.000 ε, ε, νέους οι οποίοι δεν έχουν καταρτιστεί και δεν έχουν απασχόληση και μπόρεσαν να χρησιμοποιήσουν τους πόρους αυτού του ταμείου. Πρόκειται για ένα, έχει έναν προϋπολογισμό 500 εκατομμύρια, παρόλα αυτά όμως, παρά το γεγονός ότι η δράση του Ταμείου είναι δράση ουσίας, έχουμε να κάνουμε με ένα πολυσχηδές σχήμα, γι' αυτό είναι δύσκολο να λειτουργήσει έμπρακτα. Η πρόταση έγινε ε, δεκτή από το Κοινοβούλιο γενικά, υπήρξε δηλαδή ευρεία συνένεση για να εργαστούμε πάνω σε αυτή την πρόταση που προήλθε από εσάς. Όμως το κατόφλι ήταν πολύ σημαντικό, το κατόφλι εργαζομένων. Εσείς προτείνατε ένα κατόφλι, εμείς μιλήσαμε για 200 εργαζόμενους, όχι της ίδιας επιχείρησης. Αποκλειστικά, 200 λοιπόν ε, επιλέξιμοι εργαζόμενοι και επίσης θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η ενεργειακή μετάβαση, οι τεχνολογικές αλλαγές και η οικολογική μετάβαση, καθώς και η συγχρηματοδότηση που θα πρέπει να είναι ένα ουσιαστικό στο στοιχείο, καθώς και η πολυτομεακή και πολυπεριφερειακή διάσταση. Όλα αυτά για να βελτιώσουμε τη δράση αυτού του Ταμείου το οποίο θα πρέπει να φέρει το όνομα Ταμείο Μετάβασης πλέον. Μέσα στα πλαίσια του Ταμείου θα υποβάλω μία τροπολογία αύριο στην Ολομέλεια γιατί θα πρέπει να βοηθούμε τους εργαζομένους στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης αλλά είναι ουσιώδες να λάβουμε υπόψη ότι υπάρχουν κερδισμένοι από την παγκοσμιοποίηση αλλά και πολύ χαμένοι. Αυτό αφορά και περιφέρειες που έχουν υψηλό δίκτυ ανεργίας ή χαμηλό δίκτυ απασχόλησης ή επιχειρήσεις που έχουν υποστεί πολλές αναδιαρθρώσεις, γι' αυτό θα πρέπει οι τοπικοί παράγοντες να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αυτό το μεγάλο τραύμα της αναδιάρθρωσης για να ενισχύσουμε την στρατηγική, την εδαφική μας στρατηγική. Η Caterpillar στο Βέλγιο, στο Σαρλερουά, έκανε πυρήνες ε, αναδιάρθρωσης για να συνοδεύσει τους εργαζόμενους να βρουν μια άλλη εργασία, αλλά και έναν άλλο πυρήνα, πυρήνα ονόματι Catch, που, είναι, που αφορά μάλλον τις επιχειρήσεις, τα πανεπιστήμια και τους τοπικούς παράγοντες για την αναδιάρθρωση και τη νέα απασχόληση, την εξέβρεση εργασίας των εργαζομένων που έχασαν την απασχόλησή τους. Άρα αύριο θα ζητήσω, θα υποβάλω μάλλον αυτή την τροπολογία, γιατί πολλές φορές είναι δύσκολο να πείσω τους συναδέλφους να τη δεχτούν για να λάβουμε φυσικά υπόψη την εδαφική διάσταση. Υπάρχουν περιφέρειες πλούσιες ή άλλες εγκαταλειμμένες και δεν μπορούμε να αφήσουμε τους εργαζόμενους μόνους σε αυτή την κατάσταση απογοήτευσης. Ελπίζω να με υποστηρίξουν οι διάφορες δυνάμεις και να, οι διάφορες ομάδες, συγγνώμη, και να υποστηρίξουν αυτή την τροπολογία. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα το λόγο έχει η Επίτροπος Τίσεν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητέ Πρόεδρε, μέλη από το 2007 το Ταμείο Αντιμετώπισης της Παγκοσμιοποίησης δείχνει την αλληλεγγύη του στους εργαζόμενους που έχουν χάσει την εργασία τους λόγω παγκοσμιοποίησης ή της ε, παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης. Έχουμε ήδη δώσει 631 εκατομμύρια ευρώ για 150 ε, επιχειρήσεις και 150.000 εργαζομένους που έχουν πληγεί τα τελευταία χρόνια. Αλλά τα πράγματα έχουν αλλάξει ε, τότε και γι' αυτό θα πρέπει να αναπροσαρμόσουμε το Ταμείο και τον κανονισμό του με βάση τα νέα οικονομικά πλαίσια. Χαίρομαι για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μας υποστήριξε για το νέο κανονισμό για το επόμενο πολιετές και επίσης τη μείωση του κατοφλίου που είχαμε προτείνει. Ε, ευχαριστώ την Μαρία Αρένε και όλους ε, τους βουλευτές της Επιτροπής Απασχόλησης και βεβαίως σας ευχαριστώ και για τη σπουδή με την οποία προχωρήσατε το Κοινοβούλιο υποστηρίζει, μάλλον υποβάλλει πολλές τροπολογίες, δέχομαι μερικές από αυτές που διασαφηνίζουν το κείμενό μας. Άλλες, σε άλλες τροπολογίες ε, έχουμε πολλές ανησυχίες και επιφυλάξεις. Ένα από τα βασικά στοιχεία της πρότασης ήταν η διαδικασία επιτάχυνσης της κινητοποίησης και θα πρέπει να έχουμε την ίδια και αν εισαγάγουμε την ίδια διαδικασία κινητοποίησης θα απεραντολογούμε και δεν θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε αυτούς τους εργαζόμενους που έχουν χάσει την εργασία τους ε, τάχιστα. Επίσης, ε, μιλήσαμε για μείωση του κατοφλίου και επέκταση της ε, περίοδου αναφοράς. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι το Ταμείο επηρεάζεται από τις απολύσεις που ήδη γίνονται Εάν φτάσουμε στους 250 εργαζόμενους, δηλαδή από τους 250 στους 200, τότε δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτούς τους μεγάλους κλειδονισμούς και δεν θα δείξουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί προστιθέμενη αξία με βάση τον, τον κανονισμό αυτό. Πάντως προσμένω αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχει τώρα η συζήτηση με ομιλητές από τις τέσσερις επιτροπές Διεθνούς Εμπορίου, Ελέγχου του Προεπολογισμού, Περιφερειακής Ανάπτυξης και Δικαιωμάτων των Γυναικών. Θα ήθελα ομιλητές να παραμείνουν στο χρόνο που έχει οριστεί και να μην τον υπερβαίνουν, γιατί θα θέλαμε να τελειώσουμε πριν από τις 12 τα μεσάνυχτα σήμερα. Η κυρία Γκράσβάιντερ Χάινς έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι κυρίες και κύριοι. Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχουμε τέτοιους μηχανισμούς για την προστασία των εργαζομένων. Ε, ε, άρα δεν αποφελούνται όλοι από το εμπόριο. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση έχει στόχο να υποστηρίξει εκείνου του εργαζόμενου, άνδρε και γυναίκε, που χάνουν την εργασία του λόγω τη παγκοσμιοποίηση, τη απελευθέρωση του εμπορίου ή τη τεχνολογική ανάπτυξη. Τι μα δείχνει η πραγματικότητα, ότι υπάρχουν πάντα και νικητέ και ετοιμένοι μεταξύ των κρατών μελών, των περιφερειών και της κοινωνίας ε, δεν ε, είναι ίσα μερασμένοι οι νικητές. Άρα έχουμε αυτό το ταμείο το οποίο έχει βοηθήσει πάνω από 140.000 απολυμένους από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επειδή όμως δεν απορροφάται πλήρως, πρέπει να ε, απλουστεύσουμε τις διαδικασίες, να υποστηρίζουμε τα κράτη-μέλη στην υποβολή των αιτήσεων και να έχουμε κριτήρια πιο ελαστικά και πιο διευρυμένα. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα Εκ μέρου ε, τη Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού, ο κ. Σπυρίνσκι. Πρόεδρε, τα κύρια σημεία από πλευρά τη Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού. Πρώτον, θα πρέπει ιδιαίτερα να στηριζόμαστε σε μέτρα τα οποία θα βοηθούν ε, τι πιο μειονεκτού ομάδε, τα κράτη-μέλη και τι περιφέρειε που έχουν πληγεί περισσότερο και όπου οι εθνικέ και περιφερειακές αρχέ δεν διαθέτουν επαρκεί πόρου για να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα. Οπότε η πάψη της, της λειτουργίας αφορά μια κερδοφόρη επιχείρηση. Θα πρέπει τα μέτρα να αποσκοπούν στην επανένταξη κοινωνικό κυρίως επίπεδο των εργαζομένων και Τρίτον, εάν ε, πρόκειται να δώσει με την έμεση διαχείριση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη βοήθεια, θα πρέπει να ορίσει με τρόπο διαφανή τον αρμόδιο, το τρίτο κοινό μέρος το οποίο θα αναλάβει την έμεση διαχείριση. Και βεβαίω οι εμπλεκόμενοι φορεί, μεταξύ των οποίων και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα πρέπει να σε θέση να συμμετάσχουν σε επιλογέ αυτέ. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ και εγώ. Εκ μέρου τη Περιφερειακή Επιτροπή, ο κύριο Σταμά Στόιτς. Πρόεδρε, κύριε Επιτροπέ. Η Επιτροπή μας έχει τοποθετηθεί και θα ήθελα να, ορίσω, να περιγράψω και εγώ τρεις στόχους. Καταρχάς, στις ε, οριακές τιμές από 250 πρέπει να πάμε στους 150 και να διευρύνουμε τον κύκλο των εργαζομένων που δεν έχουν απολυθεί αλλά θα μπορούσαν να απολυθούν και τρίτον θα πρέπει οι προθεσμίες να είναι στο δυνατόν πιο σύντομες. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και θα αποτέλεσε ένα πολύ μεγάλο βήμα. Πρέπει να μειωθεί λοιπόν η οριακή τιμή ως στα 150 άτομα, γιατί αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις σπάνια έχουν 500 ή 250 εργαζομένους. Δεν φτάνουν λοιπόν σε ένα κράτο μέλο ποτέ στο επίπεδο των 250 εργαζομένων. Γι' αυτό θέλουμε να μειωθεί ο αριθμό των εργαζομένων που χάνουν την ε, θέση εργασία. Ευχαριστώ και εκ μέρου τη Επιτροπή των Γυναικών η κυρία Μπλίνκεβιτσούτε. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Το Ταμείο για την Παγκοσμιοποίηση, 10 χρόνια που λειτουργεί τώρα, έχει βοηθήσει ιδιαίτερα ανθρώπους που έχουν χάσει τη δουλειά του λόγω ε, απολύς, ε, έχουν χάσει την εργασία του λόγω της παγκοσμιοποίησης. Πρέπει να βελτιωθεί με το νέο ταμείο η στήριξη προς τους εργαζομένους έτσι ώστε να έχουν ταχύτερη πρόσβαση στην ε, βοήθεια πιο αποτελεσματική και με προαγωγή των, της ισότιμης μεταχείρισης των φύλων. Είναι σοβαρό το χάσμα και η διαφορά μεταξύ των φύλων ε, στα θέματα που έχουν να κάνουν με τα μαθηματικά ή με την πληροφορική. Έτσι λοιπόν θα μπορούσαμε να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στην κατάρτιση των γυναικών για τους τομείς αυτούς όταν έχουν χάσει τη θέση εργασία τους για να καλύψουν αυτό, αυτή την υστέρηση σχέση με τους άντρες που μάλιστα έχουν και καλύτερες αμοιβέ. Πρέπει λοιπόν οι γυναίκες που αναζητούν μια θέση εργασίας ή που μπαίνουν σε κατάρτιση επαγγελματική να εξασφαλίζουν την κατάλληλη υποστήριξη ε, σε όρους απτούς. Ε, σας ευχαριστώ πολύ ο Πρόεδρος. εργασία η που μπαινουν σε καταρτιση επαγγελματικη να εξασφαλιζουν την καταλληλη υποστηριξη σε ορους τους. Σα ευχαριστω πολυ ο προεδρος και ετσι ολοκληρωνουμε τον καταλογο των ομιλητων που εκπροσωπουν κοινοβουλευτικε επιτροπε και τωρα περνουμε στου ομιλητε εκ μερου των πολιτικων ομαδων πρωτη η ομαδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο με τον κύριο Φάντεν Κεντελάρα. Έχετε το λόγο. Κύριε Επίτροπε, συνάδελφοι, το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Παγκοσμιοποίηση απέθανε τουλάχιστον από το 2021 θα γίνεται λόγος για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Μετάβασης, όχι προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση αρχικά ε, ε, ε, πρόκειται, για ένα ταμείο που βοηθούσε τους ανθρώπους που έχαναν τη δουλειά τους από τις προσαρμογές και τις μεταρρυθμίσεις. Και θυμούνται όλοι τη Φόρτ στην πόλη της Φλάνδρας ή την Caterpillar που ακούσαμε προηγουμένως στο Σαλερουά. Τώρα έχουμε μια εκβάθρονα αναθεώρηση του Ταμείου. Και ευχαριστώ Ρητά και συγχαίρω την Επίτροπο για την πρότασή της δεν είχε σχεδιαστεί καλά το ε, εργαλείο αυτό το ταμείο και γι' αυτό δεν είχε πλήρη απορρόφηση. Ήταν πάρα πολύ στενό το πεδίο εφαρμογή και τώρα το διευρύνουμε στην ψηφιοποίηση και στην αυτοματοποίηση. Και επίση ε, το κατόφλι των εργαζομένων. 250 ε, εργαζόμενοι είναι πολλοί, αλλά πολλοί είναι και 150 γιατί υπάρχουν περιοχέ αραιοκατοικημένε που χρειάζονται ιδιαίτερη κατάρτιση και μετεκπαίδευση εργαζόμενοι. Καταφέραμε ως Κοινοβούλιο ε, να μειώσουμε το 250 στο 200. Αλλά θέλουμε να μειώσουμε πολύ και το γραφειοκρατικό κόστος και το διοικητικό. Είναι λογικό ότι ένας απολυμένος θέλει πολύ γρήγορα να ξαναβρει δουλειά. Ε, δεν χρειάζεται μια μεγάλη ανάλυση για το τι έγινε και γιατί έχασε τη δουλειά του. Ε, και με το Brexit 28.000 θέσεις εργασίας θα ανοίξουν στη δική μου περιφέρεια από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Υπάρχει λοιπόν πολύ μεγάλη ε, δουλειά ακόμα να γίνει. Ευχαριστώ από τους σοσιαλιστές και δημοκράτες η κυρία Άχνες Γιονχέριους. Πρόεδρε, όταν σε μια περιφέρεια της Ευρώπης απολύονται πολλοί άνθρωποι ταυτόχρονα, αυτό αποτελεί μεγάλο πλήγμα για όλη την περιφέρεια. Και όταν έχουμε έκτακτες περιστάσεις θα πρέπει να μπορούν οι άνθρωποι να υπολογίζουν γρήγορα στην υποστήριξη και την αλληλεγγύη της Ευρώπης. Γνωρίζουμε ότι αλλάζει η εργασία, οι μορφές εργασίας με όλες τις τεχνολογικές εξελίξεις, με το διεθνή ανταγωνισμό, με την παγκοσμιοποίηση και θα πρέπει και εμείς να προσαρμοστούμε και στην κλιματική αλλαγή γιατί και αυτό θα έχει επιπτώσει στην αγορά εργασίας. Οι άνθρωποι που πλήττονται από αυτές τις αλλαγές δεν θα πρέπει να εγκαταλείπονται στη μοίρα τους και εγκαίρως να φροντίσουμε να ε, βρουν δουλειά, να μπορούν να υπολογίζουν στη δική μας υποστήριξη και στη στήριξη για να μπορούν να ε, ξαναβρούν δουλειά. Γι' αυτό υπερψηφίστε αυτό το Ευρωπαϊκό Ταμείο ε, Μετάβασης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και ε, μας, δώσατε, μας χαρίσατε δύο δευτερόλεπτα. κύριος Χότς από το ΙΣΙΑ. Ευρωπαϊκή Φούντου το 2007 Το Ταμείο για την Παγκοσμιοποίηση συστήθηκε το 2007. Χρειάζεται λοιπόν τώρα να βελτιωθεί, να γίνει πιο αποτελεσματικό, να υποστηρίζει καλύτερα τους εργαζόμενους που χάνουν τη θέση εργασίας τους λόγω της παγκοσμιοποίησης. Οι εργαζόμενοι λοιπόν στο μέλλον θα μπορούν να την χάνουν υποστήριξη εάν, είναι, εάν η θέση εργασίας τους μετατράψει και σε ψηφιοποιημένη, μηχανοποιημένη ή, σε, ή λόγω της παγκοσμιοποίησης. Πρέπει να περιορίσουμε λοιπόν τον αριθμό των εργαζομένων σε 100 στους 150, να μειώσουμε την γραφειοκρατία, να βελτιώσουμε τη σχέση μεταξύ μικρότερων και μεγαλύτερων επιχειρήσεων που δεν έχουν μέχρι τώρα αξιοποιήσει μεγαλύτερων και μικρότερων που δεν έχουμε μέχρι τώρα αξιοποιήσει το μέσο. Επτά μόνο χώρε το έχουν αξιοποιήσει. Είναι ενδιαφέρον να κοιτάξει κανεί και τα ποσά. 68 εκατομμύρια Ιρλανδία, 100 εκατομμύρια η Γαλλία, η Ελλάδα, η Δανία, το Βέλγιο, ελάχιστα εκατομμύρια, ούτε ένα εκατομμύριο άλλη χώρα. Στην Πολωνία, παραδείγματι, γιατί δεν χρησιμοποίησαν το ταμείο αυτό προηγουμένες κυβερνήσεις με 4.000 ναυπηγούς, ε, εργάτες των ναυπηγείων ε, που έκλεισαν και που ε, είχαν απολυθεί. Ευχαριστώ. Άλντε. Κυρία Φέκκα πέρα. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Αρχικά το Ταμείο για την Παγκοσμιοποίηση είχε συσταθεί για την ε, προσφορά υποστήριξης στους εργαζομένους που έχασαν λόγω της παγκοσμιοποίησης τη θέση εργασίας τους. Επέτρεπε στους ε, ανθρώπους αυτούς να βρουν μια νέα θέση εργασίας ή κατάρτιση, νέα κατάρτιση και νέες δεξιότητες. Ωστόσο, πλέον ε, η ανεργία δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι οφείλεται μόνο στην παγκοσμιοποίηση, αυτοματοποίηση, ψηφιοποίηση, προξενούν πιέσει για αλλαγέ σε πολλού τομεί τη οικονομία και πολλοί είναι αυτοί που φοβούνται ότι θα χάσουν τι εργασίε του. Ε, το νέο λοιπόν αυτό το ταμείο. Το Ταμείο Μετάβαση είναι πολύ πιο ευέλικτο, επιτρέπει την αντίδραση σε αυτέ τι μεγάλε προκλήσει και την προετοιμασία των εργαζομένων έτσι ώστε να προσαρμοστούν καλύτερα στι νέε συνθήκε. Είναι πολλέ οι αλλαγέ που έχει επιφέρει στο Ταμείο η Επιτροπή αλλάζει ο χαρακτήρας του Ταμείου αυτού και ως εκ τούτου πρέπει να είμαστε κάπως επιφυλακτικοί στο γεγονός, παραδείγμα ότι είχαμε το όριο των 500 απολύσεων μέχρι τώρα. Η Επιτροπή θέλει να τις μειώσει στις 250, ενώ το Κοινοβούλιο ζητάει ακόμα λιγότερες, 200 απολύσεις για να ενεργοποιηθεί το Ταμείο. Είναι πολύ σημαντικό όμως για τους εργαζομένους των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, γιατί αν αυτές ε, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιμετωπίσουν κρίση. Η κρίση επηρεάζει ολόκληρες περιφέρειες χωρί όμω να πρέπει να είναι και τα κριτήρια υπερβολικά χαλαρά. Γιατί αν περνούμε σε όλο και μικρότερε επιχειρήσει για τη χορήγηση βοήθεια, το... ο κίνδυνο δεν είναι το ταμείο αυτό να αφεμαχθεί, να ζητούνται συνέχεια δηλαδή ποσά από αυτό και τελικά να μην ε, προστατεύονται επαρκώς οι εργαζόμενοι ή αλλιώς να επιβαρυνθεί ιδιαίτερα η γραφειοκρατία. Επίσης το Ταμείο θα πρέπει να περιορίζεται σε απρόβλεπτες εξελίξεις, στην κάλυψη συνεπειών απρόβλεπτων εξελίξεων, και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και το Brexit βεβαίως, το οποίο είναι μια τεράστια διευθυντική αλλαγή. Σημαντική όσο και οποιαδήποτε άλλη στην Ευρώπη. Πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι θα χάσουν τη θέση εργασία του λόγω του Brexit. Ευχαριστώ πολύ. Πράσινη η Μόνικα Βάνα. Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε, αξιότιμοι συνάδελφοι, αξιότιμες συνάδελφοι. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Παγκοσμιοποίηση με, ανα, αλλάζει όνομα και γίνεται Ευρωπαϊκό Ταμείο Μετάβασης. Εμείς ως Πράσινη ζητήσαμε την, ε, είχαμε κάνει την πρόταση αυτή για να είναι δυνατή η έκφραση της ισότιμης μεταχείρισης των καλών θέσεων εργασίας, της υποστήριξης για τη μετάβαση. Είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για την πολιτική ε, την κοινωνική για τα εργατικά, για να μπορεί να προστατευτεί ο εργαζόμενος, τον οποίο δεν προστατεύουν πολλά μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι λοιπόν τη κοινωνική Ευρώπη στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Μετάβαση. Χαίρομαι ιδιαίτερω διότι η κοινή μα εργασία έχει επιτρέψει αρκετέ βελτιώσει. Βελτιώσει που περιμένουμε να δούμε υλοποιούνται στο μέλλον. Αφενό μεν στρέφεται προ το μέλλον. Αναφέρεται στην ψηφιοποίηση αλλά και την μετάλλαξη της ε, κοινωνίας που εγκαταλείπει της ε, παραγωγής της οικονομίας η οποία ε, εγκαταλείπει σιγά σιγά τον άνθρακα πράσινες θέσεις εργασίας Αναφέρεται επίσης στους νέους που δεν είναι ούτε στο σχολείο, ούτε εργάζονται, ούτε είναι σε κάποια μορφή κατάρτιση, στους νίτς δηλαδή, τους περιλαμβάνει και αυτούς. Έχει σημαντική βελτίωση σε σχέση με τα ποσοστά συγχρηματοδότησης και παρέμβασης μειώνεται ο αριθμός των προστατευομένων ατόμων, μάλλον των ατόμων για τα οποία μπορεί να χορηγηθεί η υποστήριξη. Ελπίζουμε να μπορέσει να εγκριθεί λοιπόν. Ωστόσο δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε την τροπολογία της εισηγητρίας διότι θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό τα μέσα του Ταμείου Παγκοσμιοποίησης να φτάνουν απευθεία στους εργαζόμενους και όχι να περνούν πρώτα μέσα από κάποιους θεσμικούς φορείς όπως το Κοινωνικό Ταμείο. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος και εκ μέρου της ΓκουΕ τώρα ο κύριος Πιμέντα Λόπες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεχόμαστε αρκετές από τις προτάσεις της εισηγήτριας που βελτιώνουν το κείμενο, αλλά οι βελτιώσεις δεν αποτελούν παρά ένα καταπραϊντικό στα προβλήματα των μετατοπίσεων και τη συγκέντρωσης κεφαλαίου και της εκμετάλλευσης των εργαζομένων που αποτελούν φτηνό εργατικό δυναμικό. Μιλάμε για χιλιάδες εργαζόμενους που στην Πορτογαλία, για παράδειγμα, έχασαν την εργασία τους. Αυτό είναι ευθύνη των πολυεθνικών. Πιστεύω ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις θα πρέπει να αναλάβουν το κόστος ε, ανάληψης νέας εργασίας, εξέβρεσης νέας εργασίας από τους εργαζόμενους και πρωτίστως να παραμένουν στη θέση εργασίας τους. Ευχαριστώ πολύ από το EFTD. Ο Τζόναθαν Άρνοτ έχει το λόγο. Οι τροπολογίες 97 και 98 μιλούν για τις επιπτώσεις της απόσυρσης του, και του Brexit δηλαδή, της απόσυσης του Ηνωμένου Βασιλείου. Και βλέπουμε ότι η Τερίζα Μέη έχασε, είναι η μεγαλύτερη ήττα στην ιστορία των Τόρις. Ελπίζω όμως να είχαμε να κάνουμε με μία αξιόπιστη συμφωνία. Δεν ξέρω λοιπόν εγώ τι να κάνω ως προς αυτό το ταμείο. Αν αλλάξουμε το όνομα δεν αλλάζουμε την ουσία Μιλάμε για περίοδο 21-27 και αυτό δεν έχει πλέον ίσο σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο, γιατί δεν ξέρουμε τι θα συμβεί και στο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρουμε τι θα συμβεί μετά το Brexit και στην περίοδο 21-27. Γιατί τη στιγμή που αντιδημοκρατικές δυνάμεις δρούν στο Ηνωμένο Βασίλειο, δεν ξέρω τι πρέπει να πω. Στην ουσία γίνεται χρήση των χρημάτων των φορολογουμένων που στην ουσία πληρώνουν για τη μελλοντική απόσυρση, αλλά θα πρέπει να κάνουμε στη συνέχεια αιτήσει για να ανακτήσουμε αυτά τα χρήματα. Νομίζω ότι το, το ίδιο το Ταμείο και η λειτουργία του αποτελούν ένα μεγάλο λάθος. Ο, ο κύριος Κάζα έχει το λόγο. Η Ευρώπη θα πρέπει να υποστηρίξει τους εργαζόμενους όταν χάνουν την εργασία τους. Αυτά τα μέτρα είναι στρατηγικής φύσης, μακροχρόνια. Αλλά θεωρώ ότι το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση λειτουργεί πολλές φορές διαφορετικά. Είναι ένα ουσιαστικό ταμείο το οποίο χρησιμοποιείται υπό συνθήκες τις οποίες δεν μπορούμε να προβλέψουμε. Δεν είναι ένα τακτικό ταμείο δηλαδή. Χρησιμοποιείται για τους απολυμένους, για τους άνεργους λόγω οικονομικής κρίσης. Βλέπω πως ερφαμόζεται και δεν συμφωνώ καθόλου με τον ε, προλαλήσαντα. Ξέρω πως έχει χρησιμοποιηθεί μέχρι τούδε, γιατί οι απολυμμένοι ακολούθησαν μια διαδικασία κατάρτισης και μπόρεσαν να εργαστούν σε νεοσύστατες εταιρείε. Θα πρέπει όμως να ξαναδούμε το όριο των ε, απολυμμένων, δηλαδή θα πρέπει να μιλάμε για ένα κατόφλι από 500 σε 250 εργαζόμενους για να μπορούμε να αντικατοπτρίζουμε τη... και τα μεγέθη των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα για μικρές χώρες όπως η Μάλτα. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μπρεσόχη το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, ε, δυστυχώς η παγκοσμιοποίηση οδήγησε σε αρνητικά αποτελέσματα. Γι' αυτό η Ευρώπη θα πρέπει να προστατεύσει τους ίδιους τους πολίτες από αυτό τον αρνητικό αντίκτυπο, να μπορέσει λοιπόν να προωθήσει την βιώσιμη ανάπτυξη για να μην υπάρχει αθέμητος ανταγωνισμός. Θα ήθελα να τονίσω τη σημασία αυτού του Ταμείου που βοήθησε περιφέρειες που αντιμετώπισαν μεγάλες δυσκολίες. Θεωρώ ότι θα πρέπει να μειώσουμε το κατόφλι για την ενεργοποίηση του Ταμείου και να λάβουμε υπόψη περισσότερες επιχειρήσεις, γιατί έχουμε να κάνουμε με μικρότητες οντότητες οι οποίες δεν είχαν ληφθεί υπόψη. Δεν μπορούμε να λάβουμε υπόψη μόνο τη διάσταση, δηλαδή η διάσταση των περιφερειών έχει σχέση και με τη διάσταση της κρίσης σε αυτές. Θα πρέπει αυτό το ταμείο να είναι ένα ταμείο οικολογικής μετάβασης και μέσα στα πλαίσια της βιώσιμης ανάπτυξης. Σε αυτή την περίπτωση οι εργαζόμενοι θα πρέπει να είναι στο επίκεντρο ενός νέου συστήματος ανάπτυξης. Τώρα το λόγο έχει η κυρία Ζαβοβιέτσκα. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Χαίρομαι γιατί έχουν ε, επέλθει αλλαγές για το Ταμείο Αντιμετώπισης της Παγκοσμιοποίησης για την περίοδο 21-27. Έτσι λαμβάνουμε υπόψη τις ανάγκες της ευρωπαϊκής οικονομίας και των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μόνο τις μαζικές απολύσεις, αλλά να δούμε κατά πόσο υπάρχει αυτοματοποίηση και ψηφιοποίηση που μειώνουν τις ε, θέσεις εργασίας. Ένα τέτοιο ταμείο θα πρέπει να συνεργάζεται με το ECT Θεωρούμε ότι πολλές εργασίες χάνονται λόγω της ε, αυτοματοποίησης και θα πρέπει να λάβει υπόψη αυτή την πρόκληση το Ταμείο. Οι άλλες αλλαγές είναι σκόπιμες ιδιαίτερα της ε, ΜΜΕ και τη μείωση του κατοφλίου από 500 ή 250, ακόμα και 200 εργαζόμενους, όπως όρισε η Επίτροπη Απασχόλησης. Θα ήθελα να πω στην κυρία Χάρκιν ότι οι εργαζόμενοι οι οποίοι χάνουν τις, τη θέση τους λόγω Brexit θα πρέπει να υποστηριχθούν. Σας ευχαριστώ πολύ. Μιχάλη Ντέτχεν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε τίποτα δεν είναι τόσο σταθερό όσο η αλλαγή. Σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία ταξιδεύουν ε, σε όλη την Ιφίλιο και καθίστανται επιχειρήσεις. Έχουμε λοιπόν εδώ νικητές και χαμένους. Αυτό που θέλουμε εμεί να εξασφαλίσουμε είναι όταν έχουμε μαζικέ απολύσει και αναδιαθρώσει, οι άνθρωποι, οι επιχειρήσει, οι κλάδοι και οι περιφέρειε να προστατεύονται και να βοηθούνται οι άνθρωποι να βρουν δουλειά. Γι' αυτό το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Κοσμιοποίηση έχει σημαντική συνεισφορά. και ελευθερώνει κονδύλια ε, για απολύσει άνω των 200 ατόμων, που δίνουν νέε προοπτικέ στου ανθρώπου και του βοηθούν να αντισταθμίσουν κάπω τι απώλειε. Ε, ε, παίζει ρόλο και η οικονομία και η παγκοσμιοποίηση, η ψηφιοποίηση, η αυτοματοποίηση και μπορεί κάπως να αυλυνθεί η επιρροή τους με τη βοήθεια του ταμείου αυτού στο μέλλον θα πρέπει να ε, συμβιώνουν αρμονικά η οικονομία, η οικολογία και τα κοινωνικά ζητήματα προς όφελος των ανθρώπων. Ευχαριστώ η κυρία Βερόνικα Λόπε Φοντανιέ, παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρία Επιτροπέ, το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βοήθεια ε, για την Παγκοσμιοποίηση έχει απεδειχθεί ε, πολύ αποτελεσματικό για τους απολυμμένους που έχασαν τη δουλειά τους λόγω της παγκοσμιοποίησης. Καταφέραμε να το προσαρμόσουμε και τώρα το προσαρμόζουμε ξανά για να συμπεριλάβουμε την αυτοματοποίηση και την ψηφιοποίηση. τεχνολογική αλλαγή ε, αλλάζει συνεχώς τις διαδικασίες παραγωγής και εμείς θα πρέπει να προσέχουμε έτσι ώστε οι πολιτικές μας να προσαρμόζονται στην πραγματικότητα. Από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συνεχίσουμε να επενδύουμε στους ανθρώπους και να βελτιώνουμε τις δεξιότητες τους γιατί μιλάμε για μεγάλους αριθμούς πολλές φορές απολυμένων. Γι' αυτό θεωρώ σημαντικό το Ταμείο αυτό να διατηρήσει το χαρακτήρα που έχει, να μπορεί να αντιδρά στις καταστάσεις και συμφωνώ και με τη μείωση ε, των οριακών τιμών έτσι ώστε να ε, κινητοποιείται νωρίτερα σε, με λιγότερους εργαζομένους έτσι αυτό προσαρμόζεται στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα ε, όπου είναι τέτοιο ο ιστό της παραγωγής και τη βιομηχανία ώστε οι μαζικέ απολύσει να αφορούν κάθε φορά και λιγότερου εργαζομένου. Ευχαριστώ. Ο κύριος ε, Σάιμον. Ε, Κύριε Πρόεδρε, παίρνω το λόγο. Μία ώρα μόλις και ακριβώς αφότου με άνευ προηγουμένου πλειοψηφία ε, ψήφισε η Βρετανική Βουλή των κοινοτήτων να καταψηφίσει το σχέδιο για το Brexit της Τερέζα Μέιν. Και συζητούμε για ένα ταμείο που θα διαθέτει κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, σε περιοχές όπου έχουν πληγεί από την ενεργεία κάποιοι. Εγώ μιλώ εκ μέρους των Δυτικών Midlands του Ηνωμένου Βασιλείου. Είναι περιοχές αυτές όπου λόγω της ψηφιοποίησης, ε, λόγω της εργασίας σε πλατφόρμες κτλ. Ε, πολλές θέσεις εργασίας χάνονται. Την προηγούμενη εβδομάδα η Jaguar και Land Rover ε, ε, ανακοίνωσε ότι θα απολύσει 4.500 εργαζομένους. Και δυστυχώς αυτό το ταμείο δεν θα ωφελήσει εργαζομένους του Ρωμένου Βασιλείου. Ούτε τώρα ούτε ποτέ. Σας ευχαριστώ πολύ για την τοποθέτηση αυτή που μας βάζει σε σκέψεις. Κύριε Λέναρς. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Στην Ευρώπη ε, το θέμα δεν είναι μόνο τα χρήματα, η αγορά και το νόμισμα, αλλά είναι και οι άνθρωποι οι άνθρωποι που ζουν ε, κάποιε κρίσει και χάνουν τη δουλειά του, απολύονται λόγω τη παγκοσμιοποίηση, θα πρέπει να του βοηθήσουμε να βρουν καινούργια θέσει εργασία. Αυτά δεν είναι αριθμοί και αφηρημένε στρατι... στατιστικέ. Είναι ε, άνθρωποι που μένουν στην Ολλανδία, στη... δεν βρίσκουν δουλειά στη Φριζία ή είναι στην περιοχή Χέλτερλαντ ε, που χάνουν τη δουλειά του γιατί κλείνουν οι τράπεζε. Άνθρωποι που ζουν κοντά στα σύνορα. Είναι πραγματικοί αληθινοί άνθρωποι με αληθινά προβλήματα. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να σκέφτεται μόνο τι επιχειρήσει, αλλά και του ανθρώπου που δουλεύουν σε αυτέ και να ψάχνει λύσει. Αυτό ακριβώ κάνει το Ταμείο παγκοσμιοποίηση και με τρόπο αποτελεσματικό και επιτυχή. Σήμερα λοιπόν θα πρέπει να στείλουμε και εμεί ένα μήνυμα και τα επόμενα χρόνια θέλουμε να βοηθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση τους ανθρώπους που χρειάζονται ε, μια στήριξη για να προχωρήσουν στη ζωή τους. Ευχαριστώ πολύ. κυρία Ρωμάνα Τόμς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχει παρέλθει μια δεκαετία από την ε, θέσπιση του Ταμείου Υποκοσμοποίησης. Πολλές αλλαγές έχουν λάβει χώρα εντωμεταξύ και γι' αυτό και ήταν σκόπιμο να αλλάξουν οι κανόνες λειτουργίας του. Πρέπει να είναι πιο απλή, με νέα κριτήρια, να καλύπτουν περισσότερους δικαιούχους ιδιαίτερα να απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στα κράτη-μέλη. Ωστόσο, πρέπει να είμαστε πιο φιλόδοξοι, πιστεύω, για το ε, όριο, για το κατόφλι. Γιατί με βάση τα στατιστικά δεδομένα στη χώρα μου, μόνο 350 επιχειρήσεις θα πληρούσαν τα νέα αυτά κριτήρια των 250 εργαζομένων. Με τις αλλαγές αυτές οι εργαζόμενοι οι οποίοι λόγω της ψηφιοποίησης και των νέων τεχνολογικών πρόοδων χάνουν την θέση εργασίας τους θα μπορούσαν να υποστηριχθούν. Πρέπει να είναι οι κανόνες λοιπόν στο δυνατόν πιο απλοί αλλά βέβαια να ελέγχεται η λειτουργία του Ταμείου. Ευχαριστώ πολύ και έτσι ολοκληρώνεται ο κατάλογος των ομιλητών. Περνώ στη διαδικασία Catch the Eye. Ο κύριος Χωσέ Φαριάν είναι πρώτος στον καταλογό μου, δεν τον βλέπω στην αίθουσα. Η κυρία Σόιντροβα, λοιπόν, παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι. Το σχέδιο τροποποίησης του κανονισμού για το Ταμείο για την Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση με βρίσκουν ε, σύμφωνοι, ιδιαίτερα όσον αφορά τη μείωση του ορίου των εργαζομένων και την παράταση της προθεσμίας. Πρέπει να κοιτάξουμε και από την ε, οπτική γωνία των, μικρότερων ε, κρατών, όπως η Τσεχική Δημοκρατία, τι αντίκτυπο μπορεί να έχει. Και γι' αυτό θα ήθελα και πιο απλοποιημένες διαδικασίες για τα κράτη-μέλη για τη διαχείριση των αιτήσεων και βέβαια από την Επιτροπή πρέπει να γίνεται η διεκπαιρέωση σε ταχύτερο χρονικό διάστημα. Χαίρομαι που το Κοινοβούλιο προτείνει την χρηματοδότηση κινήτρων για τους εργοδότες για τις θέσεις εργασίας ε, μερικής απασχόλησης που θα βοηθούσαν ιδιαίτερα γονείς ε, να επανέλθουν στο χώρο εργασίας. Κύριος Μαριάς, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, συζητούμε το Ταμείο για την αντιμετώπιση των συνεπειών της παγκοσμιοποίησης νομίζω ότι έχει αποδείξει ότι πραγματικά προσέφερε στήριξε τους εργαζομένους σε μια φάση όπου είχαμε μαζικές απολύσεις. θα έλεγα βέβαια για την περίπτωση της ελλάδος ότι δεν αξιοποιήθηκε τόσο πολύ όσο μπορούσε διότι φαίνεται και από τα κονδύλια τα οποία διατέθηκαν στην ελλάδα τα οποία ήταν πολύ λίγα σε σχέση με το συνολικό ποσό το οποίο διατέθηκε. σε κάθε περίπτωση είναι ένα ταμείο το οποίο μπορεί να στηρίξει τις περιφέρειες να στηρίξει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να δώσει τη δυνατότητα μετάβασης και στο πλαίσιο αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσει πλέον και τις συνέπειες της αυτοματοποίησης επομένως ε, τα μέτρα τα οποία προτείνονται στο βαθμό που απευθύνονται καθαρά για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και κυρίως για τη στήριξη των ίδιων των ανέργων είναι πάρα πολύ θετικά. το ότι πρέπει το κατόφλι να κατέβει στους 200 εργαζόμενους από 500 που ήταν πριν επίσης το θεωρώ πολύ σημαντικό. ας εξετάσουμε να φτάσει το κατόφλι και στους 150 εργαζόμενους. ευχαριστώ.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 η παγκοσμιοποίηση έχει μεγάλη ε, σημασία και μεγάλο αντίκτυπο στις ε, περιφέρειες μας, στο Βίγκο, την πόλη μου, αλλά και στη Γαλλικία και στην Κορούνια. Επίσης, μας έπληξε η παγκοσμιοποίηση και δεν ξέρουμε τι θα γίνει με την Αλκόα στην ε, Κορούνια και στην Αβιλές. Ξέρετε ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι το Ταμείο δεν εφαρμόστηκε με διαφάνεια και θα θέλαμε η Επιτροπή να επαγρυπνεί στην ε, εφαρμογή του Ταμείου, τη διαφάνεια, τη ε, συμμετοχή των συνδικάτων, όπως είδαμε τη συνέβη στη Γαλλική από την ε, τοπική κυβέρνηση. Αυτό είναι ένα θέμα ύψης της σημασίας. Δυστυχώς, οι πολλές επιχειρήσεις δεν έγιναν ε, δεκτές γιατί δεν υπήρχε συμμόρφωση με, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας του κράτου μέλους. Στάνισλαφ Πόλτσακ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να υποστηρίξω αυτό το μέσο. Πιστεύω ότι είναι ιδιαίτερα ευεργετικό για τις ε, περιφέρειες που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση ή έχουν πληγεί από την παγκοσμιοποίηση. Βοηθά επίσης και τις βιομηχανίες που έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση. Εξ αρχής θεώρησα το Ταμείο ένα εξαιρετικό μέσο εάν εστιάζαμε την προσοχή μας σε αυτό το βασικό ζήτημα της απώλειας θέσεων εργασίας θα είχαμε αποφύγει ίσως και το ίδιο το Brexit. Θα ήθελα να πω ότι αυτά είναι ζητήματα που είναι ύψης της σημασίας όπως είπε και ο εκπρόσωπος του Ηνωμένου Βασιλείου. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι είναι ένα ποιοτικό μέσο για τους πολίτες. Η Επίτροπος Τίσεν έχει το λόγο. Για να ολοκληρώσει τη συζήτηση. Thank you, Mr. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη και πάλι καλωσορίζω το γεγονός ότι θα εγκρίνει την πρότασή μας στο Κοινοβούλιο σε πρώτη ήδη ανάγνωση. Και χαίρομαι για τις επόμενες ε, συζητήσεις. Ε, αυτό τι δείχνει, ότι η έκθεση του Κοινοβουλίου ε, θα αποτελέσει τα γερά θεμέλια για τις διοργανικές διαπραγματεύσεις που θα ακολουθήσουν. Όπως πάντα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πρόθυμη να γίνουν συζητήσεις στον τριμερή διάλογο και θα διαδραματίσουμε το ρόλο μας ως έντιμος μεσολαβητής. Με την αναθεώρηση αυτής ε, της νομοθεσίας δεσμευτήκαμε να δώσουμε στο Ευρωπαϊκό Ταμείο για την ε, παγκοσμιοποίηση το χώρο και το ρόλο που ε, του ανήκει. Χαίρομαι που συμφωνείτε με αυτές τις πρωτοβουλίες και ελπίζω να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των πολιτών. Θέλω να ευχαριστήσω και πάλι το Κοινοβούλιο για την πάγια υποστήριξή του και την ταχεία έγκριση και είμαι πεπισμένη ότι κατά τη διάρκεια της Ρουμανικής Προεδρίας θα φτάσουμε σε μία πρώτη γενική ε, συμφωνία. Ε, αυτά θα τα συζητήσει το Μάρτιο η ε, Επιτροπή ΕΠΣΚΟ το, το Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ, λέει ο Πρόεδρος. Ε, ευχαριστώ την κυρία Επίτροπο και γενικά για τη συζήτηση. Ε, κλείνει η συζήτηση. Η ψηφοφορία θα γίνει αύριο. Α. Επόμενο θέμα στην μέρη της διάταξη. Α, όχι, κάνω λάθος, λέει ο Πρόεδρος. Η κυρία Μαρία Ρενά έχει το λόγο, η συγγήτρια. Ευχαριστώ, κύριε πρόεδρε. Καταρχά, θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ανέλαβε αυτή την πρωτοβουλία, γιατί χωρί την νομοθετική πρωτοβουλία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήταν δύσκολο εμεί να εργαστούμε για να βελτιώσουμε το Ταμείο. Ευχαριστώ την Επιτροπή και όλε τι ομάδε και του κοιόδη ηγητέ. Ε, συνεργαστήκαμε για την νέα νομοθεσία αυτή και πάλι θα του ζητήσω να κάνουν ακόμα μια προσπάθεια κατά τη διάρκεια της ψηφοφορία αύριο. Δηλαδή, όταν εμείς εργαζόμαστε για την πλαισίωση των εργαζομένων, είναι πολύ σημαντικό να μιλούμε και για την κατάρτιση. Αλλά αν μετά την κατάρτιση δεν δημιουργούνται θέσεις εργασίας ε, για τους ανθρώπους αυτούς, ε, είναι δύσκολο να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να περάσει η τροπολογία που προτείνω αύριο για να υπάρχει και αυτό το αντιστάθμισμα. Θα πρέπει να προχωρούμε και να πατάμε σε δύο πόδια. Από τη μια να εκπαιδεύουμε και να καταρτίζουμε τους εργαζομένους μας, αλλά από την άλλη έχουμε και επιχειρήσεις που να ανοίγουν δουλειέ για να μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να ξαναμπούν στην αγορά εργασίας. Ελπίζω να υποστηρίξουν όλες οι πολιτικές ομάδες που υποστήριξαν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Μετάβασης. Ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστώ. Κυρία εισηγήτρια, με συγχωρείτε για το ατόπιμα. Το διόρθωσα όμως. Ολοκληρώνεται εδώ η συζήτηση, ψηφοφορία αύριο. Και τώρα αγαπητοί συνάδελφοι, περνάμε στο επόμενο θέμα της μέρης της διάταξης. Εκθέση Βερόνα Καλόπη Φοντανιέ για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Plus. Και πάλι θα λάβουν το λόγο μετά την εισηγήτρια εκπρόσωποι των κοινοβουλευτικών επιτροπών και μετά θα γίνει συζήτηση. Ξεκινούμε με την εισηγήτρια. Βερόνικα Φοντανή. παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, πριν να αρχίσω με την παρέμβασή μου, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους, επόμε... τους ε, άλλους κοιόδες για την εξαιρετική συνεργασία κατά τις διαπραγματεύσεις, αλλά θα αναφερθώ και αργότερα σε αυτούς. Το κείμενο της Επιτροπής ήταν ε, μεγάλη βοήθεια γιατί υπάρχουν διάφορα ταμεία μέσα στα πλαίσια του ΕΕΚΤ και αυτό θα βοηθήσει στην άρση των διοικητικών προσκομμάτων και την απλούστευση. Επίσης, η σύνδεση με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο θα επιτρέπει στα κράτη-μέλη να επικεντρώσουν την προσοχή στα πιο σημαντικά για αυτά σημεία. Αυτό θα πρέπει να είναι στο επίκεντρο των πολιτικών μας. Βεβαίως, η οικονομική ανάκαμψη είναι δεδομένο, αλλά έχουμε μεγάλο δρόμο μπροστά μας. Θα πρέπει να αυξήσουμε την εργασία των νέων, να βελτιώσουμε τα εκπαιδευτικά συστήματα, προσαρμόζοντάς τα στην αγορά εργασίας, επίσης να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε τους εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας και να μειώσουμε την κοινωνική φτώχεια. Αυξάνεται σε 27% η χρηματοδότηση του ΕΚΤ συν έτσι ώστε να φτάσουμε σε ειδικέ αντιμετώπιση ειδικών ομάδων όπως η Ρωμά. Επίσης 3% επιπλέον για τις ε, ε, ομάδες που μειονεκτούν, καθώς και συνοδευτικά μέτρα για την ε, βοήθεια συμμετοχής αυτών των ομάδων. Επίσης, βοήθεια προς τους νέους για να μπορέσουν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Αυτό είναι προτεραιότητα για μας. Θα θέλαμε όλα τα κράτη-μέλη να προσδίνουν το 3% των πόρων για τους ε, νέους που δεν έχουν εργασία και εκείνους που ε, θα πρέπει να έχουν μία εργασία. Ε, δηλαδή να προσδώσουμε ένα 15%. Ένα 24,5% των ανηλίκων βρίσκονται σε κατάσταση κινδύνου και κοινωνικού αποκλεισμού. Πρόκειται για απαράδεκτους ε, δείκτες. Η φτώχεια των ανηλίκων αποτελεί ένα θέμα κοινωνικής συμμετοχής. Αν θέλουμε όλοι οι πολίτες να έχουν ίσες ευκαιρίες, θα πρέπει να εργαστούμε από την παιδική ηλικία. Γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε 5,9 δις για την εντετόπιση της παιδικής φτώχειας. Η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών έχει μεγάλη σημασία. Το άρθρο 6 αναφέρεται στους πρωταρχικούς όρους και κάνει λόγο για ειδικέ ε, δράσεις για τη συμμετοχή των γυναικών. Επίσης, τα άτομα με αναπηρία θα πρέπει να μπορούν να συμμετέχουν στο κοινωνικό γίγνεσθε όπως ορίζουν και τα Ηνωμένα Έθνη και θα πρέπει φυσικά να υπάρχει και πρόσβαση στην εκπαίδευση και την εργασία. Και τέλος θα ήθελα να μιλήσω για την κοινωνική οικονομία, γιατί γίνεται λόγος για έναν επιμερισμό, για μεγαλύτερη νομική ασφάλεια και θα βοηθήσει και άλλες επιχειρήσεις σε χώρες όπως Ιταλία, Ισπανία και Πορτογαλία, όπου το ε, ΕΚΤ ασχολείται με τους πολίτες που είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Όντως, είναι μια έκθεση με μεγάλο φάσμα. Οκτώ είναι οι επιτροπές που έχουν γνωμοδοτήσει, περιβάλλον, προπολογισμός, έλεγχος του προπολογισμού, περιφερειακή ανάπτυξη, εκπαίδευση, πολιτισμός, ε, πολιτικές ελευθερίες γυναικών. Και έτσι ξεκινούμε με την πρώτη, με τον πρώτο μιλητή εκ μέρους Επιτροπής Περιβάλλοντος. Ο κύριο Μπουσόη, παρακαλώ. Θα ήθελα να λάβουμε υπόψη ότι είχαμε τρία προγράμματα στον τομέα της υγείας που είχαν πολύ θετικά αποτελέσματα στην Ρουμανία. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τι μπορεί να κάνει το ΕΚΤΣΙΝ. Στον τομέα και της υγείας, η ΕΜΒΗ ζήτησε ένα ξεχωριστό πρόγραμμα για την υγεία, γιατί η υγεία αποτελεί προτεραιότητα με βάση και το τελευταίο ευρωβαρόμετρο, διότι η πλειοψηφία των πολιτών θέλουν μεγαλύτερη παρέμβαση στον τομέα της υγείας. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχουν σαφείς στόχοι που να τηρούνται. Η Επιτροπή Περιβάλλοντος μίλησε για τον τομέα της υγείας ιδιαίτερα και μιλήσαμε για 473 εκατομμύρια ευρώ μέσα στα πλαίσια της ε, βιώσιμης ανάπτυξης για την πρόληψη ε, ασθενειών και έγινε λόγος και για τη δημιουργία μιας διευθυντικής επιτροπής για να δούμε ποιες είναι οι συνέργειες με άλλα προγράμματα στον τομέα της υγείας πάντα. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Τίσεν έχει το λόγο.